δεν, έχει, δεν είναι σε θέση να συζητήσει το νέο ε, σύνταγμα της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ πολύ. La parola quindi alla commissaria... Το λόγο λοιπόν έχει η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ.